<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. Καλημέρα σα. Κυρίσω την έναρξη τη συνεδρίασή μα. Okay, okay, start. Witam Państwa bardzo serdecznie. Σα καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίασή μας. και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες πριν την ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έχουμε μία αλλαγή. Η ψηφοφορία για το σημείο 4, τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών, αναβάλλεται για την επόμενη μας συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 26 Απριλίου. Τότε θα ψηφίσουμε. Αυτό μας ζήτησε η συγγύτρια η κυρία Μακιντάιρ, την αναβολή της ε, ψηφοφορίας, γιατί είχε επίγουσες ε, υποχρεώσεις στην πατρίδα της, στην Αγγλία. Γι' αυτό και αναβάλουμε την ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση, της 26 Απριλίου. Τώρα, για το τη διερμηνίας έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσε. με εξαίρεση αισθανικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών 20 ε, Δευτέρα και 23 Φεβρουαρίου και 7 η Μαρτίου, ε, ισχύει η κανονική διαδικασία μέχρι το τέλο συνεδρίας. Παρακαλώ παρατηρήσει. Και περνάμε στο σημείο 5, την ενίσχυση τη καινοτομία και τη οικονομική ανάπτυξη στην ε, μελλοντική διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Ο κύριος Χαΐτεμα είναι η εισηγητής μας. Έγινε ήδη η ανταλλαγή απόψεων ε, και μάλιστα 300 και τροπολογίε κατατέθηκαν για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και μάλιστα αυτέ τι 312 τροπολογίε δείχνουν το ζωηρό ενδιαφέρον που προκαλεί αυτό το θέμα της ενίσχυσης της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος. Αλλά αυτό το θέμα είναι σημαντικό για το σύνολο του γεωργικού τομέα. Πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός του κλάδου, ανανέωση, προκειμένου να έχουμε υψηλότερες προδιαγραφές και καινοτομίας. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους και οδησηγητές γιατί κατέληξαν σε μερικές συμβαστικές τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε την ψηφοφορία. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Χέιτεμα, παρακαλώ. Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους και οδησηγητές των πολιτικών ομάδων για την πολύ καρποφόρα συνεργασία που είχαμε και καταφέραμε να ε, περιλάβουμε πολλές τροπολογίες και να τις ε, ομαδοποιήσουμε και να τις συγχωνεύσουμε σε συμβιβαστικές. Πολύ σημαντικό θέμα, η καινοτομία και οι νέες προτάσεις για να βελτιωθεί η οικονομική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, αλλά να βελτιωθεί και ο αντίκτυπος ε, στο περιβάλλον, αλλά και να βελτιωθεί η μεταχείριση των ζώων. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τη συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή και ευελπιστώ ότι η έκθεσή μου θα συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία. Και εμείς το πιστεύουμε και το ελπίζουμε κύριε Ισηγητά. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Περνάμε στην Τροπολογία 102, διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 102, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία 102. Τροπολογία 98. Ποιος είναι υπέρ της 98? Ε, μόνο. Πρώτα την τροπολογία 101 όμω γιατί η 102 είχε απορριφθεί. Ποιο είναι υπέρ τη 101? Εγκρίνεται, ωραία. 98 τώρα, ποιο είναι υπέρ? Εγκρίνεται, ευχαριστώ. Συμβαστική τροπολογία Α. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ως συνήθως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία Β. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 118. Ποιος είναι υπέρ της 118. Κατά. Απορρίπτεται. 120. Ποιος είναι υπέρ. Διανατάσεις της χειρός παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 17 προς 18 παρατρίχα. Απορρίπτεται. Εκατόν επανάληψη, γιατί η κυρία Μαγκίνες δεν πρόλαβε να ψηφίσει. Ή όχι, δεν χρειάζεται. Α, καλά, εντάξει. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως. Αν ήσασταν υπέρ θα άλλαζε το ποτέ. Αλλά ούτως ή άλλως και υπέρ να ήσασταν πάλι ισοπαλία οδηγεί στην απόρριψη. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις για κανέναν. Α, είστε και αντιπρόεδρος. 122. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σε, σι, Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία σε γάμα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 124. 124 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της 124. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία R. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε, τροπολογία 11 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 11 MV. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατα... Ε, εγκρίνεται. Τροπολογίες 132 και 133 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κύριε Ντές, 132 και 133 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, λέω. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 136. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. απορρίπτονται. 137. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 137 κατά. Απορρίπτεται. 139. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 140. Ποιος είναι υπέρ της 140. Κατά. Απορρίπτεται. 142. Ποιος είναι υπέρ της 142. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά απορρίπτεται 147 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται 148 ποιος είναι υπέρ Εγκρίνεται. 151. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 152. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. D. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία ΔΕΛΤΑ. Τέλος. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 164. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 24 της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος υπέρ κατά απορρίπτεται. 166. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 167. Πάνω μειότυπη. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πάμε στην 168. ή μάλλον 170. 170 ποιος είναι υπέρ του κυρίου Ντόρφμαν. Εγκρίνεται. 172. Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν και νομίζω ότι είχε απορριφθεί 172. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 172 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. 174. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 175 υπέρ. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Ο Απορρίπτεται. 180. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 182 υπέρ εγκρίνεται. 183 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική σύγματα Υπάρχει πρόβλημα τεχνικό. Άρχεται λέει η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία F. Α, έχουμε πρόβλημα τεχνικό. Εντάξει, διορθώθηκε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική Πάμε στην τροπολογία 5 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 188. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 189. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη. 195 πρώτα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Δικιά σου τροπολογία ψήφισε. Κατά. Απορρίπτεται. 190. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Εγκρίνεται. 193 υπέρ. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Εγκρίνεται. 197 ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 202 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Εγκρίνεται και αυτό. 203. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 208. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί. 211. Ή μάλλον 210. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αρρύπτεται 213 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για τη 213 άρχεται η ψηφοφορία Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Przyjęta. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 221. Στην τροπολογία, συγγνώμη, 221. Ποιος είναι υπέρ της 221. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 226. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 227 υπέρ εγκρίνεται 228 υπέρ εγκρίνεται 229 υπέρ εγκρίνεται 230 υπέρ κατά απορρίπτεται 231 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία J. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία J. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 259. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 259 εγκρίνεται. 258 και 261 μαζί παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 262 και 260 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 263 υπέρ κατά απορρίπτεται 264 υπέρ απορρίπτεται 265 υπέρ εγκρίνεται 267 υπέρ κατά απορρίπτεται 268 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο έχει καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την τροπολογία 268. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 273. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 273. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν είχα καλή ορατότητα. Πάμε στη 270. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. 271 υπέρ. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 272 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 274. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 275. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 277 του κυρίου Δεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 280. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 278. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 279. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία κάπα Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμβη 10 τώρα. Τροπολογία 10 της Έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 288 και 289 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες 288 και 289. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος. Απορρίπτονται. Τροπολογία 287. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 294 υπέρ κατά απορρίπτεται 293 υπέρ κατά απορρίπτεται 290 Σρέιερ πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ εγκρίνεται και αυτό 291. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 292. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Η 90 είχε απορριφθεί. 13. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία L. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στην 304. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 307. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Εγκρίνεται. 305. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. 305. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 312 εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 2 και 3 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 4 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία μη Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, έρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ, 13 και 14 μαζί. Είναι πανομοιότυπες. Κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 18 και 16 παρομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 19 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα όμως για τις δύο προηγούμενες τροπολογίες 18 και 16 άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie. Sprawdzamy elektronicznie. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Τέλος. εγκρίνονται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Εγκρίνεται. 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 και 32 ταυτόσιμες. Μαζί λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. 33 και 31 παρόμοιες υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 34 υπέρ, εγκρίνεται. 35 υπέρ, εγκρίνεται. 36 και 37 παρόμοιες επίσης. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Ελεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 36 και 37 έρχεται ψηφοφορία. Κάμι 36 Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Σας το είχα πει εγώ. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ο μικρόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας Przechodzimy, przyjęta. Przechodzimy do Πάμε στην 64 τροπολογία. Εγκρίθηκε η προηγούμενη συμβαστική. Ποιο είναι υπέρ τη 64. Εγκρίνεται. 66 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π. Άρχεται ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη τροπολογία 80. 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Q. Άρχεται ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική Q. Πάμε στην 90. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 90. Εγκρίνεται. 89. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογίες 88, 92 και 93 είναι παρόμοιες. Ψηφίζουμε μαζί ποιος είναι υπέρ των τριών τροπολογιών. Κατά απορρίπτονται. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, χαλάλη σας Ηλεκτρονικό έλεγχο για τις τροπολογίες 88, 92 και 93 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 94. Ποιος είναι υπέρ. 94. Κατά. Απορρίπτεται. 97. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Και τώρα ολόκληρο το σχέδιο ψηφίσματος όπως έχει τραποποιηθεί. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλο τη Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία της έκθεσης Χόιτεμα. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά και συγχαρητήρια και στους συνεργάτες σας. Μήπως ε, θέλετε κύριε Σιγητά, κύριε Γιάν Χόιτεμα, μήπως θέλετε το λόγο. Σας είπαμε τα συγχαρητήρια, μήπως θέλετε το λόγο. Μεγάλη μου χαρά για την ευρεία στήριξη της έκθεσης αυτής και είναι και πολύ καλό για τη σημασία που έχει η έκθεση και το θέμα της. Σίγουρα είναι σημαντικό το θέμα, αλλά και δύσκολο ταυτόχρονα. Περνάμε στο σημείο 6. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόσφατη αποστολή της Επιτροπής Γεωργίας στις κάτω χώρες. 29 με 31 Μαρτίου 2016. Όπως ξέρετε, ε, αμέσως μετά τις ε, πασχαλινές διακοπές, μία αντιπροσωπεία μας μετέβη στην Ολλανδία με τον υποφαινόμενο πρόεδρο. Επικεφαλής αντιπροσωπείας. Ε, θέμα ήταν η καινοτομία, η τεχνολογία στην Γεωργία, αλλά και θέματα περιβαλλοντικών επιδόσεων, καλής μεταχείρισης των ζώων και ανταγωνιστικότητα. Είδαμε λοιπόν επί τόπου ε, καινοτόμες ε, δράσεις στην γεωργία, όπως είναι ένα φυτό που βοηθά στην εξαγωγή και ανάκτηση, ανάπτυξη φωσφορούχου άλατος από τα λοιπάσματα προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί. Είδαμε λοιπόν ε, στην πράξη αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή μας ε, και οργανωτή της ε, επίσκεψης, τον κύριο Χαϊτεμα. Θα του δώσω σε λίγο το λόγο. Η γραμματεία θα ετοιμάσει το σχέδιο έκθεσης ε, της αποστολής. Ήταν αρκετά περίπλοκα τα θέματα. Γι' αυτό χρειάζεται κάποιος χρόνο στη γραμματεία για να εκπονήσει την έκθεση. Πάντω όταν είναι έτοιμη θα σα τη μοιράσουμε. Και τώρα λόγω στον κύριο Χέιτεμα για να μα ενημερώσει για την αποστολή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που πήραν μέρος ε, στην αποστολή αυτής της κατοχώρας. Ήξερα ότι για κάποιους ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν γιατί ήταν αμέσως μετά το Πάσχα, αλλά για όσους τα κατάφεραν τους ευχαριστώ. Πραγματικά σκοπός της αποστολής ήταν να δείξει επί του πρακτέου τι κάνουμε με τις προσπάθειές μας για καινοτομία και νέες ιδέες. Κάθε νέος τομέας στην Γεωργία, κάθε διαφορετικός τομέας, η γαλακτοκομική, εντατική, οι βιολογικές καλλιέργειες, είναι μορφές που προσπαθούν να υλοποιήσουν νέες ιδέες και νέες τεχνικές για να βελτιώσουν ή να ενισχύσουν την οικονομική του ανταγωνιστικότητα και να περιορίσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στο πρόγραμμα πρώτα απ' όλα πήγαμε σε μια εταιρεία που είναι ειδικευμένη στην ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των ε, καλλιεργειών, όχι μόνο με υλικά προστασίας, προσπαθώντας να μην χρησιμοποιεί λοιπάσματα αλλά μικροοργανισμούς ή έντομα, για να μην χρησιμοποιούνται τόσα υλικά φυτοπροστασίας και με ολοκληρωμένη προστασία των σωδιών, διότι ακριβώ με του μικροοργανισμούς και τα έντομα προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση των κατασκευασμένων λιπασμάτων ή τη ε, τεχνητή κοπριάς τη ζωική μάλλον κοπριά, η οποία μόνο ε, με, φυσικά ορυκτά μπορεί να προσληφθεί πιο εύκολα και από τα ίδια τα φυτά. Ήταν ένα καλό παράδειγμα λοιπόν για το πώ η δύναμη τη φύση και το να βλέπουμε τη φύση ω ε, σύμμαχο μπορεί να μα βοηθήσει να περάσουμε και σε καινοτομία. Σε δεύτερη φάση είδαμε κάποιε εκμεταλλεύσει που ασχολούνται περισσότερο με την με τη γεωργία ακριβίας ε, με συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και τεχνικές, το οποίο, συμβαίνει, το, οποίο το χρησιμοποιούν και στα ακροκτήματα, με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, με GPS και με συστήματα άρδευσης όπου δεν χρειάζεται παρουσία ανθρώπου. Εδώ περιορίζεται πάλι η χρήση λιπασμάτων ε, και των φυσικών υλικών, διότι σημειώνουν ακριβώς τι χρειάζεται το φυτό ή το ζώο που εκτρέφεται, προτού ξεσπάσει μια νόσος ή υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Επίσης ένα ακόμη ενδιαφέρον μέρος, ότι πήγαμε σε δύο εκμεταλλεύσεις που εξειδικεύονται σε νέο σύστημα στέγασης, στάβλησης για τα ζώα και για την ευζοία τους, με συνέπεια να, χρησιμοποιείται λιγότερο, να χρησιμοποιούνται λιγότερο τα αντιβιωτικά. Αυτό το είδαμε σε βοηδή και σε νεαρά βοηδή για την παραγωγή γάλακτος. Επίσης η διαδικασία για την παρασκευή κόπρου στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας μας απασχόλησε, διότι αυτή τη στιγμή Αυτό που ισχύει πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς 170 κιλά αζότου ανά εκτάριο όπως ίσχυε τώρα με τους νέους κανόνες. Πρέπει λοιπόν οι γεωργοί να αγοράζουν τεχνητά λιπάσματα, όχι φυσική κόπρο και υπάρχουν πλέον νέες τεχνικές για να καθαρίζεται η ζωική κόπρος και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα απευθείας. Με τη νέα νομοθεσία για τα λιπάσματα Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μα για να πούμε ότι οι τεχνικέ αυτέ καλό είναι να διαδοθούν περισσότερο. Η ζωική κόπρο να αξιοποιείται ώστε τα τεχνικά, τεχνητά λοιπάσματα να περιοριστούν. Η παρασκευή τεχνητών λοιπασμάτων έχει μεγάλη, ε, μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την εκπομπή διοξιδίων αερίων του θερμοκηπίου και παράγει και φωσφορού χάλατα. Ε, εν τέλει, Συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Γεωργίας και τους προσώπους του Υπουργείου για σκοπούς ε, διαδικτύωσης και νομίζω ήταν ευχάριστο, ε, μπορώ να το πω εγώ ίδιος πιστεύω, να ε, συναντηθούμε για ένα δείπνο εργασίας σε ένα μουσείο με πολλά έργα φλαμανδών και γενικότερα άλλων μεγάλων ζωγράφων και με εκπροσώπους και του βιομηχανικού τομέα της Γεωργίας αλλά και του Υπουργείου μας. Ήταν πολύ κατάλληλη στιγμή να τους συναντήσουμε. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ να τις θέσετε, αλλά βεβαίως και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε απορίες για το θέμα αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χαίταμα. Η κυρία Σρέιερ η τωρα το λόγο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη εργασία στην Ολλανδία. Όλα όσα είδαμε ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έχω μια ερώτηση σε σας ε, Πρόεδρο. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την καινοτομία στην αγορά και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά αυτό το οποίο συζητάνε αυτή τη στιγμή στην ε, Ολλανδία και το συζητήσαμε και χτες το βράδυ με τον κλάδο έχει να κάνει με την κρίση στη γεωργία, την τιμή δηλαδή των προϊόντων. Και εδώ πέρα ακριβώς θα ήθελα ακριβώς να μεταφέρω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο τους αγρότες στην Ολλανδία και το συζητάνε κάθε μέρα στα σπίτια τους. Και βεβαίως ε, ε, οι γεωργοί θεωρούν πως χρειάζονται την Ευρώπη ακριβώς για να παρέχει λύσεις. Αυτό το βρήκα πάρα πολύ φανταστικό ε, που το είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Χάιτεμα, αλλά ως Ολλανδέζα θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται, πώς λειτουργούμε εδώ μέσα, γιατί καμιά φορά χάνω και εγώ λίγο την μπάλα. Κατά λοιπά, σας ευχαριστώ για την πολύ καλή επίσκεψη. Δύσκολα, δύσκολα αυτά. Η κυρία Γιλέρα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή αποστολή στην οποία συμμετείχα. Έμαθα πάρα πολλά για τη γεωργία ακριβίας στην Ολλανδία και τις προκλήσεις ε, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χάρη στην καινοτομία. Η Ολλανδική Γεωργία ήταν ανέκαθεν ε, σύγχρονη, πρωτοπόρος και ανταγωνιστική. Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά καταρτισμένο και νομίζω ότι όλοι μάθαμε πάρα πολλά. Και θα ήθελα να συγχαρώ όλους ιδιαίτερα στον κύριο Χαϊτεμα για την εξαιρετική διοργάνωση και να ευχαριστήσω και τους ε, συντρόφους συναδέλφους της Ολλανδικής Αντιπροσωπείας που μας συνάδευσαν, Πραγματικά ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και πολύ ικανοποιητική και απολαυστική αυτή η αποστολή. Και περιμένουμε την έκθεση τη σχετική. Πολύ καλή οργάνωση και πολύ ενδιαφέρουσα και σαφώς ευθυγραμμισμένη με τους στόχους που είχαμε θέσει. Δεν βλέπω να θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε ήρθε και η δικιά μου σειρά γιατί έλαβα και εγώ μέρος στην αποστολή. Ήταν πολύ ε, εντατικό το πρόγραμμα. Φυσικά επικράτησαν τα θέματα της καινοτομίας και της γεωργίας ακριβίας. Και ήταν πολύ θετικό που στα θέματα αυτά της καινοτομίας χρησιμοποίησαμε και αξιοποίησαμε καλύτερα τα λιπάσματα και το, το πώς θα τροφοδοτούμε με λιπάσματα ε, τη γεωργία ακριβίας. Ε, ξέρετε ότι στην Ολλανδία έχουμε κατακόρυφη ολοκλήρωση Και έτσι έχουμε τα διάφορα επίπεδα της ε, μεταποίησης και του εμπορίου που συνδυάζονται με τη γεωργία και δεν ξέρουμε πού σταματάει η γεωργία και πού ξεκινάει το εμπόριο μερικές φορές. Και νομίζω ότι οι γεωργοί υποφελούνται στην Ολλανδία από κάποια συμπληρωματικά εισοδήματα χάρη σε αυτή την ολοκλήρωση που εφαρμόζεται. Άλλες χώρες ε, είναι λίγο πιο πίσω σε αυτά τα θέματα. έχουμε μεγάλο, μεγάλη συμμετοχή και του μεταπητικού τομέα και των επιχειρήσεων ε, της διοίκησης. Η φορολογία είναι αρκετά υψηλή. Ε, είδαμε καταπληκτικά τοπία και πολύ ωραίες ε, εικόνες. Δεν είδαμε και πολλούς Γεωργούς βέβαια. Αλλά οι δικοί σας Γεωργοί δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Είναι επιχειρηματίες δεν είναι η τυπική χαρακτηριστική Γιώργη. Πάντως λάβαμε πολλές πληροφορίες και από τον Προεδρεύοντα Υπουργό Γεωργίας για το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Βέβαια ακούσαμε και τα παράπονα για την κρίση του γαλακτοκομικού τομέα. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση και έχουμε και κοινή αγορά, οπότε είναι κοινά τα προβλήματα. Πάντως, πραγματικά συναντήσαμε και το φοιτητέ από το Πανεπιστήμιο Wageningen και κορυφαίο πανεπιστήμιο και νιώσαμε και εμείς μερικές φορές σαν φοιτητέ μαθαίνοντας τόσα πράγματα και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα την επιστήμη και την καινοτομία στην γεωργία ακριβίας. Κάτι που το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως, αλλά το συνειδητοποίησαμε πολύ καλύτερα σε αυτή την αποστολή. Οπότε, συμφωνώ κι εγώ και επαναλαμβάνω τα συγχαρητήρια της κυρίας Αγγιλέρα. Και τώρα, ε, Μπήκε πολύ ψηλά ο πήγης κυρία Αγγιλέρα, γιατί η επόμενη μας αποστολή θα είναι στην Ισπανία και είστε εσείς η οργανώτρια. Βέβαια στην Ισπανία είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της γεωργίας και είναι κατανοητό. κύριος Ντόρφμαν ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ σύντομα να ευχαριστήσω και εγώ τους Ολλανδούς συναδέλφους για την πάρα πολύ οργάνωση του ταξιδιού. Ένα πράγμα παρατήρησα εγώ κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού μας είπαν πως υπάρχει νομοθεσία η οποία εμποδίζει κατά κάποιον τρόπο την καινοτομία. Επισκεφτήκαμε παραδείγματο χάρη μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει καινοτόμα συστήματα, βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας και τους λένε και μας είπαν πως υπάρχει νομοθεσία η οποία τους δυσκολεύει τη ζωή γιατί η αναγνώριση ενός βακτηρίου ε, για να αντιμετωπιστεί όπως ένα χημικό μέσο φυτοπροστασίας ε, ε, διαρκεί πάρα πολύ, περνάνε χρόνια και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι βεβαίως το ευκολότερο το οποίο έχουν να κάνουν ε, είναι να αρχίσουν να εισάγουν ε, από αλλού εκτός Ευρώπης ε, αυτά τα οποία χρειάζονται. Είναι λίγο περίεργο δηλαδή αυτό το οποίο κάνει νομοθεσία. Μάλιστα. Καλή η σύστασή σας. Και έχουμε πολύ συχνά εμπειρογνώμονες από από το Πανεπιστήμιο Βάγκενίγκεν. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τους επιστήμονες αυτού του Πανεπιστημίου ειδικά. Πάντως, πολύ πετυχημένη αποστολή και σημαντικό στάδιο της Ολλανδικής Προεδρίας, γιατί διανύουμε μια χαλεπή περίοδο και σε άλλες χώρες έχουμε προβλήματα και καλό θα ήταν να ακούμε τα παράπονα των γεωργών, γιατί είναι ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση, ειδικά στη γεωργία. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο να τους ακούσουμε στις επόμενες μας επισκέψεις. Πάντως ε, και ευρωβουλευτές από άλλε επιτροπές αρχίζουν και ενδιαφέρονται και να θέτουν ερωτήσεις για την κατάσταση στη Γεωργία, κάτι που δείχνει πραγματικά πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση. Ε, φαίνεται ότι οι Γεωργοί ε, φτάνουν και σε άλλου ευρωβουλευτές από άλλε επιτροπές και δεν απευθύνονται μόνο σε εμά. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την ε, ιδιαίτερη αυτή κατάσταση και τις υψηλές προσδοκίες των γεωργών της αγροτικής κοινότητας. Δεν μπορούμε λοιπόν να απογοητεύσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τους γεωργούς. Δεν μπορούμε να τους ρίξουμε. Και μάλιστα η κατάσταση στη Γεωργία επηρεάζεται σε, μεγάλες, σε μεγάλο βαθμό από, την εξω, από εξωτερικούς παράγοντες. Ε, από την από το σχετισμό προσφοράς και ζήτησης, από την κατάσταση στη Γεωργία, Βραζιλ... της Γεωργίας στην Αργεντινή, Βραζιλία, Αυστραλία. Είναι δύσκολο να διαφυλαχθεί αυτή η παγκόσμια ισορροπία. Πολλοί λοιπόν εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν και την εσωτερική μας κατάσταση στη Γεωργία. Ολοκληρώσαμε το σημείο 6 και θα πάμε σε λίγο στο 7. Αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι έτοιμη η έκθεση της αποστολής. Κατάφερε η γραμματεία και την εκπώνησε, οπότε θα σας την δώσουμε αμέσω. Πάμε στο σημείο 7 λοιπόν τώρα, την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης. Α, συγγνώμη, ο κύριος Χαϊτεμα πρόλαβε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε και τη γραμματεία και τους βοηθούς που οργάνωσαν το ταξίδι γιατί υπήρχε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που έπρεπε να γίνει για να κυλήσει σωστά η αποστολή και να πάμε σε τόσες πολλές εκμεταλλεύσεις σε τόσο σύντομο διάστημα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. E, ευχαριστώ. Ε, διορθώσετε τη δική μου παράληψη Φυσικά, φυσικά είναι αξιέπαινη και η γραμματεία. Μερικές φορές την ξεχνάμε. Συγγνώμη, συγγνώμη που παρέλειψε τις ευχαριστήσεις και προς τη γραμματεία. Αρχίζει και ανυπομονή βέβαια. Βλέπω τον κύριο Γιάρ να κουνιέται και να αδειμονεί. Γιατί όντως φτάνουμε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Την προετοιμασία της θέσης της Επιτροπής Γεωργίας με τη γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, για την μετακλογική αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Γιάρ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπατε ήδη πως είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η σημασία αυτή βεβαίως ε, δεν ε, αντικατοπτρίζεται τόσο στον έκταση της έκθεσης. Το θέμα είναι ο προπολογισμό ε, και τα επόμενα έτη και γνωρίζετε πως η πολιτική σημαίνει και χρήση κονδυλίων. Οπότε πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Σε δύσκολους καιρούς μπορεί κανείς να πεις, αν δει κανείς τη συνολική κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν συνεχώς νέες απαιτήσει και συνεχώς ε, συζητάμε για το πώς θα πρέπει να δώσουν τα... να εκταμιευτούν τα κονδύλια. Τώρα να ευχαριστήσω και τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Είχαμε ήδη μια πρώτη συνάντηση στις 21 του προηγούμενου μηνός. Και νομίζω πως ε, έχουμε αρχίσει να καλύπτουμε κάπως μια γενική γραμμή γιατί θα πρέπει να βρούμε και μια συνεννόηση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού γιατί δεν έχει νόημα ε, πάρα πολύ αργά να προσπαθήσουμε ως Επιτροπή Γεωργίας να επηρεάσουμε την Επιτροπή Προϋπολογισμού και να περιμένουμε να γίνουν αυτά δεκτά πρέπει να αρχίσουμε από τώρα τις επαφές. Ε, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνάντηση στις 21 Μαρτίου. 29 ε, Τετάρτου 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τροπολογίες ε, και συμφωνήσαμε όπως είπαμε 12 Μαΐου να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο και αν πάνε όλα ε, σύμφωνα με το σχέδιο 6 Ιουλίου στην Ολομέλεια πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είχαμε λοιπόν τις πρώτες ιδέες των ε, συναδέλφων και καταλήξαμε σε μια γενική κατεύθυνση. Η πρώτη αρχή στην οποία υπάρχει νομίζω μια συμφωνία είναι πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε για τον προπολογισμό. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Εμείς είπαμε όμως ότι θα παραμείνουμε στο θέμα μας. Θα μείνουμε στη συζήτηση για τον ε, προϋπολογισμό Ναι, έπρεπε βέβαια να περιοριστούμε όπως είπαμε σε αυτές τις πέντε σελίδες, ε, δεν έχουμε περισσότερο περιθώριο, απλά για να ξεκαθαρίσουμε στους συναδέλφους ε, του προπολογισμού ποιο είναι το θέμα. Αλλά όπως είπα δεν ε, έχουμε πολλά μπλα μπλα. Το βασικό λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα έλεγα μια σταθεροποίηση του προϋπολογισμού. Έχουμε λοιπόν τώρα προκλήσεις ε, μπροστά μας. Ε, έχουμε προβλήματα σε αρκετά γεωργικά προϊόντα. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι απειλούνται πλέον με εξαφάνιση. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε αυτό το οποίο θέμε ως πρώτος στόχος είναι μια σταθερότητα και εξηγούμε ότι η γεωργική πολιτική είναι πάντα πολυετής και πρέπει να χαράζεται σε βάθος χρόνου και μετά λέμε το εξής με λίγα λόγια αλλά ουσιαστικά εάν η κοινωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει συνεχώς νέες απαιτήσεις ε, στους αγρότες θα πρέπει πολύ απλά να τους δώσει και τα απαραίτητα κονδύλια. Δηλαδή τους λέμε φροντίστε να κάνετε κάτι, να υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν μπορεί να έχετε μόνο απαιτήσει από τους ε, γεωργούς. Πρέπει να υπάρξει μια σταθεροποίηση όπως είπαμε. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση με τους ε, συναδέλφους ε, της Επιτροπής υπολογισμού. και οπωσδήποτε προσπαθήσαμε να τους μεταφέρουμε το κλίμα που επικρατεί στη δικιά μας την Επιτροπή και τους είπαμε πως τρία πράγματα είναι για μας ε, ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο είναι η διατήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ότι δεν πρέπει δηλαδή να μειωθεί και να πηγαίνουν τα κονδύλια σε άλλους τομείς ε, της ε, πολιτικής, γιατί έχει αναλάβει για κάποιες νομικές υποχρεώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θέλουμε οι άμεσες πληρωμές στον τίτλο 2 να παραμείνουν ίδιες. Και αυτό βεβαίως παίζει μεγάλο ρόλο. και να μην μειωθούν και εδώ οι πληρωμές. Διαπιστώνουμε επίσης ξεκάθαρα πως ε, πρέπει να διαπιστώσουμε πως τα ανώτατα όρια τα οποία έχουν καθοριστεί για την ΚΑΠ από τον ε, προϋπολογισμό έχουμε ελάχιστο πλέον περιθώριο ελιγμών. Και θέλω να παρακαλέσω τους συναδελφούς να βοηθήσουν για να ξεκαθαρίσουμε στους συναδέλφους ε, των άλλων ε, επιτροπών ότι ε, βλέπουμε ξανά το παιχνίδι που είχαμε πριν από 10-15 χρόνια ότι τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να βρουν ένα-δύο δισεκατομμύρια από τον Επίτροπο Γεωργίας και να τα στείλουν κάπου αλλού στον προπολογισμό. Αυτοί οι καιροί πλέον έχουν παρέλθει ειλικρινά Ε, τονίσαμε ποιες είναι οι ανάγκες μας ε, και μας ε, έδωσαν μετά ένα κομμάτι του προπολογισμού, αλλά πλέον δεν υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στους συναδέλφους. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε το πρόβλημα ότι οι νέες προκλήσεις αυτές είναι μεγάλες. Έχουμε το μεγάλο κίνδυνο των τιμών, που ανέφερα. Έχουμε το θέμα το φυτοϊγειονομικό και της υγείας ε, των ζώων. Όλα αυτά θα μπορούσαν να επιβαρύνουν ε, τα αποθεματικά πάρα πολύ γρήγορα. Και ακριβώ λέμε στους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμού πως ε, για αν χρειαστούν λεφτά για νέα επιπρόσθετα μέτρα ανάγκης δεν υπάρχουν πλέον άλλα διαθέσιμα. Όλα αυτά λοιπόν όπως είπα φαίνονται σε 19 σημεία και ε, θα ήθελα ακριβώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Θα καθοριστούν ε, οριστικά όπως είπα στις συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και ε, Βεβαίω, όπω είπα, θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσουμε γέρο. και να συμφωνήσουμε, νομίζω, όπω συμφωνούμε, σε μεγάλο βαθμό εντό τη Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Και πριν να περάσουμε στη συζήτηση, να σας πω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε μια δημόσια κρόση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Να το ξέρουμε γιατί θα γίνει, θα γίνει η συζήτηση και χαίρομαι που είχα λάβει μέρος σε αυτή τη δημόσια κρόση της Επιτροπής Προϋπολογισμών γιατί πρέπει να ακούγεται και η φωνή της Γεωργίας. Μάλιστα, ε, διαπίστωσα ότι ένας από τους ε, ε, εμπειρογνώμονες χαρακτήρισε την Επιτροπή Γεωργία γαλακτοφόρα για Ελλάδα, για Ελλάδα για άρμεγμα. Και όσο εφαρμόζεται κοινή γεωργική πολιτική, μας λέει θα απαιτεί όλο και μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Φανταστείτε τι ε, γνώμη έχουν μερικοί εμπειρογνώμονες για την κοινή γεωρική πολιτική. Όπως ε, θα φαντάζεστε βέβαια, έλαβα το λόγο, δεν μπορούσα να κρατηθώ και μίλησα πολύ ε, ρητά και φθαρσός. Προσπάθησα βέβαια να κρατήσω την ψυχραιμία μου, αλλά ε, αγανάκτησα με το χαρακτηρισμό αυτό της κοινής γεωρικής πολιτικής. Αυτό είναι τρομερό να υπάρχει τέτοια εντύπωση. Με εξόργησε πολύ αυτή η αντιμετώπιση της Γεωργίας. Βέβαια, ήμουν ευγενικό στην απάντηση, παρόλο που μίλησα με πυγμή. Αλλά ε, μου ήρθε να τον πνίξω, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, κρατήσαμε ένα επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να έχουμε τα μάτια μας 14 για το τι γίνεται στις διάφορες επιτροπές και να επισημάνουμε το πρόβλημα και στις άλλες επιτροπές. Και να πούμε στους γεωργούς μας ε, τα προβλήματά τους να τα ανακοινώνουν στους ε, ευρωβουλευτές, όχι μόνο στις Επιτροπές Γεωργίας, αλλά και στους υπόλοιπους. Ο κύριος Αλμπερντές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε αυτά τα ζητήματα πάντα προσέχουμε και ακούμε και στη δικιά μου τη χώρα υπάρχει αυτή η διαίρεση των ειδικών και εμεί έχουμε ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα και το λέω και το επαναλαμβάνω ξανά για να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Εάν όλες οι δημόσιες δαπάνες έκαναν αυτό το οποίο κάνει η γεωργία στις ε, Βρυξέλλες τότε θα ήταν ένα εκατό και τίποτα παραπάνω. Γιατί, κοιτάξτε, η άμυνα, η παιδεία, η υγεία, όλα αυτά δεν χρηματοδοτούνται μέσω των Βρυξελών. Ενώ η γεωργία χρηματοδοτείται μέσω των Βρυξελών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν είχε... Ε, 9 ε, και 6 κράτη-μέλη τότε η ΕΟΚ ήδη ε, περνούσαν οι πληρωμές από εδώ πέρα και 1% δημόσιες δαπάνες για ε, να παρέχουμε τρόφιμα σε μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό και δεν πρέπει να, να ακούμε αυτά τα οποία λένε για 38% του προπολογισμού κτλ. Είναι ελάχιστα τα ποσά για 40 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη που φροντίζουν κάθε μέρα για το να έχουν οι καταναλωτές μας ε, ποιοτικά και επαρκή τρόφιμα. Και αυτά είναι πάντα προ όφελο του καταναλωτή γιατί τι γίνεται, είναι πιο φτηνό το τελικό προϊόν το οποίο είναι το τρόφιμο. Αυτό είχα να πω εγώ για τη χρηματοδότηση της Γεωργίας. Κύριε Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, Πέτερ Γιάρ για την έκθεση αυτή. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφο που ανέφερε πράγματι αυτό το 1% το οποίο αντιστοιχεί στον ε, προϋπολογισμό των ε, κρατών μελών. Μιλάμε για 32 cent που δίνει κάθε Ευρωπαίος πολίτης την ημέρα για να έχει επαρκή και ποιοτικά τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν εγώ θεωρώ να απαιτήσουμε ε, να μην μειωθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός. Ήδη έχει μειωθεί αρκετά και τώρα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον άλλο περιθώριο. Για μένα σημαντικό το σημείο 11, γιατί πρέπει να τονίζουμε πάντα ξεκάθαρα πως ε, χρειαζόμαστε τις αγροτικές επιδοτήσεις, έχουν, είναι άμεσες πληρωμές, ένα εισόδημα για τους αγρότες που περνάνε δύσκολες στιγμές, περνάνε μια κρίση και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και σημαντικό για εμένα επίσης είναι το σημείο 17 όπου ε, λέμε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Γιατί έχουμε την αίσθηση το ότι η γεωργική πολιτική δεν ε, λειτουργεί ακριβώς. Η λύση δεν είναι η επανεθνικοποίηση. Και το σημαντικότερο ε, για μας είναι το σημείο 19 στο τέλος όπου λέμε ξεκάθαρα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους ε, στόχους ε, μπροστά μας. Θεωρώ λοιπόν πως η τωρινή κοινή γεωργική πολιτική αυτή την οποία έχουμε τα τελευταία έτη πραγματικά δεν έχουμε μια γενική εικόνα. Τι γίνεται με το πρασίνισμα το λεγόμενο, αν είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Δεν συζητάμε λοιπόν επί της ουσίας μόνο για τα λεφτά και τον προϋπολογισμό. Και δεν ε, τίθεται το ζήτημα της κατεύθυνσης της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και το ότι ε, κατευθύνονται κονδύλια φεύγουν από τη γεωργία και πάνε στο περιβάλλον, κάτι το οποίο πρέπει να απορρίψουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά τα οποία είπατε ξεκάθαρα. Ότι δηλαδή όταν υπάρχουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις πρέπει να υπάρχουν και επιπρόσθετα κονδύλια για τη γεωργία. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Ο σκιώδη ηγητή ε, της ομάδα μου δυστυχώ απουσιάζει. Θα ήθελα όμω και εγώ να σας παρουσιάσω τη θέση τη ομάδα μου. Το σχέδιο γνωμοδότησης ε, έχει κάποια θετικά σημεία. Αναφέρεται σε κάποια βασικά στοιχεία της παρούσας ε, γεωρικής κρίσης που σοβεί στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά είναι σχετικά άτολμη έκθεση, γιατί δεν μιλά για τι πραγματικέ αιτίε τη γεωργική κρίση. Γιατί οι πραγματικέ αιτίε ε, είναι οι μεταρρυθμίσει που είναι μόνο προσανατολισμένε στην αγορά. Αναφέρεται η κρίση ω άμεση συνέπεια της καταστροφή των αρχών ε, ε, των ρυθμιστικών αρχών της προσφοράς. Κάθε φορά που έχουμε ευκαιρία, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έγινε με στόχο την απελευθέρωση του, των αγορών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, δεν αναφέρονται οι εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ε, μακροπρόθεσμε τάσεις, τάσεις μείωσης του γεωργικού εισοδήματο και ταυτόχρονα μια αυξανόμενη αστάθεια βραχυπρόθεσμη που φαίνεται στις απότομες διακοιμάνσεις των τιμών. Είναι πολύ σημαντική η γεωργία για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία που έχουν οι μικρές και μεσαίες γεωργικέ εκμεταλλεύσεις σε αντίθεση με τη βιομηχανική μεγάλης κλίμακας γεωργία, που δυστυχώ αυξάνεται και ενισχύεται χάρη στους νέους προσανατολισμού τη ΚΑΠ. Δεν λαμβάνουμε δεόντως υπόψη του στόχου της συνοχής. Είναι σοβαρότατη η κρίση στη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να ε, ζητήσουμε κάποιες δημοσιονομικές προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στην κρίση. Επίσης, ε, η υπερβολική χρήση των αποθεματικών κρίσεων εξαιτία του ρωσικού εμπάργου και ε, μετά την μείωση των τιμών που ήταν η πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία, θα πρέπει ο κοινοτικό προπολογισμό να αναλάβει τις συνέπειες αυτής της κατάστασης. Επίσης, να λύσουμε την αντίφαση μεταξύ του σημείου 6 και του 18 και να αυξήσουμε σημαντική αύξηση των κονδυλίων της ΚΑΠ, είτε στον τομέα 2, είτε στα κονδύλια των αποθεματικών της κρίσης και εκτάκτων ανάγκης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σένερα. Ο κύριος Λουαζό. Oui, merci, Monsieur Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό δυστυχώς δεν πηγαίνει παραπέρα σε πολλά θέματα, κυρίως για την ε, μείωση των ε, τιμών σε σταθερές του ευρώ από το 2000, από το που ξεκίνησε η κρίση όλος ιδιαίτερος, οπότε πρέπει να συνδεθούν οι βοηθείες χωρίς τις οποίες η απαραίτητη ανάπτυξη και η ισορροπία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας μπορεί να ε, πληγεί με δραματικά προβλήματα που προκλήθηκαν και από την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Ενώ όλε οι άλλε δυνάμει, ιδίω οι Ηνωμένε Πολιτείες, που ε, αντιμετωπίζουμε με καλύτερο τρόπο το θέμα των τιμών και των όγκων παραγωγής έχουν συγκεκριμένες διαπραγματεύσει, οι οποίες επηρεάζονται και από όσα αυτή τη στιγμή συζητιούνται στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων TTIP. Η επανεθνικοποίηση των ε, βοηθειών ε, μας δυσκολεύει με το κείμενο αυτό που δημιουργεί ένα διέξοδο με τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που ε, συνέταξε το κείμενο αυτό. Αντικατροπτίζει πιστεύω σωστά την κατάσταση όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί. Ήθελα ωστόσο και εγώ να ε, ε, εκφέρω κάποιες απόψεις. Γιατί να αυξήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα της γεωργίας και να μην τα μειώσουμε, ας πούμε. Υπόθηκε και σωστά ότι έχουμε 500 εκατομμύρια ανθρώπους να θρέψουμε στην Ευρώπη. Η γεωργία όμως η γεωργία όμως προσφέρει κάτι διαφορετικό δεν θα ήταν σωστό να συγκρίνουμε το ποσό το χρηματικό που η Ευρώπη αφιερώνει στη Γεωργία, αλλά να δούμε πώς διαβιούν οι Γεωργοί σε σχέση με τον κόσμο που ζει στα αστικά κέντρα. Λέγω χάρη στη Λιφουανία η ανεργία στην Ήπεθρο είναι διπλάσια από ότι στα αστικά κέντρα τα εισοδήματα είναι δύο φορές υψηλότερα. Χαμηλότερα μάλλον, συγγνώμη. Εάν δούμε αυτό το ποσοστό του 38% που φαίνεται υψηλό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μας λέει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το σημείο 4. Κυρίως διότι αναγνωρίζουμε ότι το κομμάτι αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, είναι μεγάλο, αλλά δεν λέει τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν... Θα ήθελα λοιπόν να διαμορφώσουμε μια σαφέστερη άποψη για την κρίση και το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Δεν δημιούργησε τα προβλήματα ο γεωργικός του κλάδος στις ε, εχθροπραξίες στην Κρυμαία ή στην ε, αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Γιατί να πληρώσει ο γεωργικός τομέας για όλα αυτά. Γιατί δεν παίρνουμε τα χρήματα και τα ποσά αυτά από τον κοινό προπολογισμό. Γιατί να πληρώσει τα σπασμένα η Γεωργία. Εάν αυτά τα κονδύλια δεν είχαμε ανακτήσει από τον κοινό προπολογισμό, μπορεί οι άλλοι να τηρούσαν πιο υπεύθυνη στάση. Επίσης, να σημειώσω ότι οι άμεσες πληρωμές είναι χαμηλότερες στις νέες χώρες. Αυτό επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα θα θέλαμε λοιπόν να εξισωθούμε με τις άλλες χώρες. Θέλουμε στην Ευρώπη να υπάρχει μια ενιαία ταχύτητα, όχι πολλές. Αλλά ο πρόεδρος θέλει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως ε, μιλήστε μετά τον κύριο Γιάρ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μιλητή. Η κυρία Γιλέρα, ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδη ηγέτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα ήθελα να πω στον κύριο Γιάρ ότι είναι σωστή η γραμμή και προσανατολισμός της γνωμοδότησης, κατά τη γνώμη μας. Γιατί μιλούμε για αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και όχι για αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν μιλούμε για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ, αλλά για το πλαίσιο, το συνολικό, δηλαδή το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό αναθεωρούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο λοιπόν. Πάντως, ε, η γενική κατεύθυνση του κυρίου Γιάρ είναι εύλογη και σωστή. Και σε αυτή την γενική προσέγγιση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και ελπίζω να υπερψηφιστεί με πλειοψηφία για να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, λόγω της μεγαλύτερης στήριξης, ώστε το, στην αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου να μην ξεχάσουμε την γεωργία και κάποια θέματα κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί χρειαζόμαστε για την κοινή γεωργική πολιτική έναν κατάλληλο προϋπολογισμό. Γιατί στον τομέα 2 όπου, όπως αναφέρεται στον κανονισμό μέχρι το 2020, στον κανονισμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, προσοχή, να μην έχουμε μείωση των κονδύλιων και να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου ε, λόγω του ρωσικού εμπάργου, λόγω της κρίσης επιμέρους τομέων και θα χρειαζόμαστε ίσως και αύξηση, όχι περικοπή του προπολογισμού. Αναφέρεται και η αστάθεια των τιμών, η υπερβολική διακύμαση. Πολύ σωστά που τα επισημαίνετε όλα αυτά. Και επίση θα πρέπει να είμαστε προορατικοί, δραστήριοι, να μην ε, παίζουμε στην άμυνα ε, είμαστε συντηρητικοί, τουλάχιστον να μην μας περικόψουν τον προϋπολογισμό. Να είμαστε πιο επιθετικοί, γιατί η ΚΑΠ εξυπηρετεί την ύπεθρο της αγροτικής περιοχές. Δεν θα πρέπει να περιμοθούν οι αγροτικές περιοχές, η ύπεθρος ε, της Ευρώπης και δεν είναι χρήματα που πηγαίνουν σε επιχειρηματίες, αλλά που ευνοούν την εδαφική συνοχή, την κοινωνική συνοχή, που βοηθούν να μην μείνουν έρημα τα χωριά και ύπεθρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση συντηρούν τα μερικά κονδύλια της ΚΑΠ τη διατήρηση της απασχόλησης σε αυτές τις ζώνες. Θα πρέπει να δείξουμε τη σημασία που έχει η ΚΑΠ επί τόπου και πόσο ενισχύει την εδαφική συνοχή. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο αμυντική στάση και να πούμε αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις στην Ευρώπη, αν μη τι άλλο να μας περικόψουν τις ΚΑΠ το, ο προϋπολογισμός ΚΑΠ δεν εξυπηρετεί μόνο κάποιου επαγγελματίε. Γι' αυτό ακόμη και θα χρειαζόταν αύξηση το προϋπολογισμό. Ο προπολογισμό τη ΚΑΠ βοηθά την ύπεθρο ε, και συμβάλλει στην εδαφική συνοχή. Αυτό το χαρακτήρα θα έχουν και οι τροπολογίε μα κυρία, και σας ευχαριστώ για την γνωμοδότησή σα. Μακάρι, μακάρι ε, να ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά ε, μερικοί σκέφτονται τα πράγματα διαφορετικά και θέλουν ακόμη και αναθεώρηση του προπολογισμού. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γιάρ για τη πολύ καλά συγκροτημένη, συστηματική και μεστή του γνωμοδότηση. Συμφωνώ ότι τα οικονομικά μέσα και κονδύλια για την κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να παραμείνουν με τι άλλο στα ίδια επίπεδα, γιατί η γεωργία συμβάλλει στον ανεφοδιασμό με τρόφιμα των Ευρωπαίων πολιτών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει και η γεωργική πολιτική στη δημιουργία ε, θέσεων απασχόλησης και σε άλλους τομείς. Ε, εφτά νέες θέσεις απασχόλησης συνδέονται με τη γεωργία κάθε φορά σε συναφείς τομείς. Γι' αυτό και θα πρέπει να δείξουμε πυγμή και να διαφυλάξουμε τον προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής και να μην μειωθεί αυτός. Ε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει χτυπηθεί από την κρίση που έπληξε και άλλους τομείς, αλλά τα μεγαλύτερα θύματα ήταν η Γεωργία μας δυστυχώς. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιάρ και να επισημάνω και κάτι που θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ε, πολλές φορές οι γεωργοί βρίσκονται στο κατόφλι της φτώχειας, ε, ειδικά όταν μπαίνουν στη σύνταξη. Μερικοί ζουν στο κατόφλι της ε, φτώχειας και μερικοί και στο κατόφλι της εξαθλίωσης όταν σταματούνται οι ορικοί τους δραστηριότητα και βγαίνουν στη σύνταξη. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε τα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν ελάχιστες γεωργικές συντάξεις. Στην ε, Κροατία έχουμε 70.000 ε, συνταξιούχους γεωργούς και η μέση σύνταξη είναι 35 ευρώ. Ποιος είναι δυνατόν να επιβεβαιώσει με 35 ευρώ το μήνα. Ποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να, να επιβιώσει με τέτοιο πενιχρό ποσό. Μην ξεχνάτε το σημαντικό ρόλο της γεωργίας και των γεωργών για μας, γιατί όχι μόνο παράγουν τρόφιμα, αλλά βοηθούν και σε πολλά άλλα θέματα. Και είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι που μας τρέφουν καθόλου τη διάρκεια της ζωής μας, αυτοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη να πεθαίνουν στην πείνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσμιουκ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ και ο να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάρ για την περίπλοκη, κατά τη γνώμη μου, γνωμοδότηση με θέμα την κοινή γεωρική πολιτική και τα φονδύλια ε, αυτής. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ταυτόχρονα και αυτό που πρόσεξε ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό ότι στην αναθεώρηση της, ε, των δημοσιονομικών προοπτικών ε, τα κονδύλια της γεωργίας ε, είναι με πολύ ελκυστικά και υπάρχει ο πειρασμός να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, όχι για την ανάπτυξη της γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε όχι μόνο την ε, διατήρηση του επίπεδου γεωργικού πολιτισμού, ε, του προπολογισμού, συγγνώμη, αλλά και την αύξησή του, γιατί χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Επίσης, ε, έχουμε μείωση των γεωργικών δαπανών απόλυτα, 75 με 80% σχέση με στο παρελθόν, και επίσης ε, πολλά γεωργικά κονδύλια κατευθύνονται σε άλλους στόχου ε, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική πολιτική, για παράδειγμα. Επίσης, εξαντλούνται τα αποθέματα εκτάκτο, ε, εκτάκτο και κρίσεων, παρόλο που αστάθεια και κρίσεις αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα σε πολλούς τομεί. Αλλά τα αποθέματα εξαντλούνται. Θα πρέπει επίσης να γεφυρώσουμε το κενό των άμεσων επενδύσεων μεταξύ παλιών και νέων χωρών. Αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές δυστυχώ ακόμη στις άμεσε ενισχύσει κοινών. ελπίζω να το περιλάβει αυτό ο κύριο Γιάννη. Ο κύριος Χόισλινγκ. <clears throat> Πρόεδρε, επιτρέψατε μου κάποιε παρατηρήσεις γιατί θεωρώ πως ε, δεν θα, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, λέμε ότι υποφέρουν οι αγρότες και χρειαζόμαστε λεφτά. Μα υποφέρουν και φουρνάριδες, υποφέρουν και άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή χρειάζεται κάποια αιτιολόγηση και θα μας πούνε στο τέλος ότι τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε για την ε, γεωργική πολιτική δεν πηγαίνουν σε αυτούς που χρειάζονται όντως τη βοήθεια και αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε τελικά εάν κάνουμε μια πολιτική συμπλήρωση εισοδήματο ή ε, ισχύει αυτό το οποίο λέμε ως αιτιολόγηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, δηλαδή ότι ε, τιμούμε την κοινωνική συνεισφορά των αγροτών. Αν είναι να τους συμπληρώνουμε το εισόδημα, θα τα βρούμε δύσκολα. Γιατί, γιατί να αιτιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, και να μην στηρίξουμε και άλλους που περνάνε κρίση και χρειάζονται λεφτά. Γιατί τα λεφτά της γεωργίας ε, πρέπει να πούμε τελικά ότι είναι λεφτά τα οποία δίνονται για κάποια πράγματα που κάνουν για την κοινωνία οι αγρότες. Και εκεί πέρα πρέπει να μείνουμε. Αυτό πρέπει να είναι το επιχείρημά μας. Οτιδήποτε άλλο δεν στέκει πάρα πολύ. Δηλαδή να ρίξουμε σε κάθε εκτάριο 300 ευρώ και να πούμε ότι είναι στήριξη εισοδήματος ε, δεν είναι το καλύτερο επιχείρημα για να υπερασπίσουμε τον προπολογισμό τη Γεωργία. Χρειαζόμαστε περισσότερα και καλύτερα επιχειρήματα. Αυτό πρέπει να, ε, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για τον προπολογισμό τη Γεωργία. αλλά να λέμε ότι όλα είναι καλά και συνεχίστε να μα δίνετε τα λεφτά γιατί έτσι τα κάναμε μέχρι τώρα, ε, δεν θα φτάσει. Το είπε και ο συνάδελφος. Υπάρχουν κρίσεις για τις οποίες χρειαζόμαστε λεφτά, όντως ε, για τις χώρες που πλήττονται από το εμπάργο, κάναμε κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτή, τη, τη βοήθεια την έκτακτη. Και το μεγαλύτερο λάθος το οποίο κάναμε νομίζω στη γεωργική πολιτική είναι ότι καταργήσαμε τους διάφορους ε, κανονισμούς ε, αγοράς, ε, π.χ. του ίνου. Όπως είπα, το αντικείμενο της ε, πολιτικής δεν μπορεί να είναι μόνο το να μοιράζουμε λεφτά. Βλέπουμε την καταστροφή στην αγορά του γάλακτος. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν είναι αρκεί μόνο να μοιράζουμε λεφτά. Πρέπει να, παρεμβούμε, να ρυθμιστικά στην αγορά. Βλέπουμε και τη ε, βοήθεια που δίνουμε στον τομέα του γάλακτος δεν φτάνουν ποτέ στους ε, ενδιαφερόμενους. Ή τι γίνεται, τα πράγματα γίνονται χειρότερα γιατί βυθίζεται ακόμη περισσότερο στο χρέος ε, το κάθε αγρόκτημα. Υπάρχει λοιπόν μάζα αγροτών η οποία υποφέρει πραγματικά και στους οποίους δεν ε, προσφέρουμε τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στην επίσκεψη εργασίας ξανά στην Ολλανδία. Είδαμε κάποιες επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, έχουν επενδύσει στην ε, καινοτομία, αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν φτάνουν στην κουζίνα τους. Ή βλέπουμε πάρα πολύ ωραία τοπία αλλά δεν βγαίνουν οι άνθρωποι οικονομικά. Ε, τα ακούσαμε και από την Rabobank ε, τα στοιχεία. 60% των ανθρώπων που εκτρέφουν ε, ε γουρούνια έχουν πρόβλημα να βγουν. Δεν αποδίδει. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Και γιατί κάνω αυτή την παρατήρηση. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, εάν το γνωρίζετε. Τι κάνουμε εμείς σε αυτή την ε, επιτροπή εδώ πέρα ασχολούμαστε καθόλου με το θέμα του περιβάλλοντος και των υπολείπων ε, υποχρεώσεων που έχουν οι αγρότες. Η Ευρώπη α, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο είχε στόχους ε, την ειρήνη και το να μπορεί να κατοικηθεί η και να καλλιεργηθεί για να έχουμε ασφάλεια διατροφική. Το θέμα αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο της δικής μας ε, επιτροπής, νομίζω πως θα έπρεπε να απασχολεί πολύ ευρύτερα ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να αφαιρθώ και σε κάτι άλλο. Πρέπει να σκεφτούμε εδώ πέρα το τι έχει αποφασιστεί στην ε, Συμφωνία για το Κλίμα. Να δούμε δηλαδή τι συνέπειες ε, θα έχει αυτό. Ίσως μπορεί να μπει την επόμενη φορά στην ημερήσια διάταξη να το συζητήσουμε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δώσω δίκιο στον συνάδελφο Χόισλινγκ, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αλλά πράγματι έχει δίκιο. Δεν είναι απλό να πούμε ότι έχουμε ένα μηχανισμό και έναν προπολογισμό και πρέπει να τα κρατήσουμε και να τα υπερασπίσουμε. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για το αν οι μηχανισμοί που έχουμε, εντάξει για τα λεφτά συμφωνώ να τα υπερασπιστούμε, αλλά οι μηχανισμοί έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί πραγματικά εξακολουθούν να είναι καλοί για μια αποτελεσματική ε, γεωργική πολιτική. Έχουμε καταργήσει διάφορα μέτρα και η γεωργική πολιτική έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα διανομής χρημάτων που συνδέεται βεβαίως με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ένα απλό σύστημα. Περισσότερα στρέμματα, περισσότερα λεφτά. Λιγότερα στρέμματα, λιγότερα λεφτά. Ή κάπως λιγότερα λεφτά. Αλλά όταν γίνουν δύσκολα τα πράγματα ή για να κάνουμε πραγματικά ουσιαστική αγροτική πολιτική δεν έχουμε πια μηχανισμούς. και θα καταλήξουμε σε πολύ δύσκολες ε, καταστάσεις ε, νομίζω και η πολιτική την οποία έχουμε αυτή την ε, στιγμή δεν ξέρω πραγματικά αν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχουμε και στην κατάσταση που έχουμε στην αγορά. Γι' αυτό ασκούμε, ακούμε ε, όλο και περισσότερη κριτική και θα ακούμε συνεχώς περισσότερη κριτική. Δηλαδή αυτά τα 50 ε, δισεκατομμύρια. Πράγματι έχει δίκιο εδώ πέρα στον Άλφο Σοντές, είναι μικρό κομμάτι του γενικού προβλήματος. τι βλέπουν οι φορολογούμενοι, τα 55 δισεκατομμύρια. Συζητάνε για τα 55 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι πράγματι πού πάνε τα λεφτά. Πάνε όντως στους ε, αγρότες και τι κάνουν. Ε, οδηγεί σε σπατάλες ή γίνονται σωστές επενδύσεις ε, στην ε, γεωργία. Ενώ βλέπουμε και μεγάλα επενδυτικά ταμεία τα οποία αγοράζουν εκτάσεις. Αυτά τα θέματα πρέπει να μπορούμε να τα απαντήσουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον προϋπολογισμό μας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Χάισλερ, ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήρθε η ώρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβουμε σύντομα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η έκθεση αντικατοπτρίζει τις βασικές μας μερίμνες, σωστά με την ενδιάμεση αναθεώρηση που αναμένεται. Είναι όμως σαφές ότι θα υπάρξει και ε, συζήτηση για τις προτεραιότητες του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι πρόσφατες γενικές εξελίξεις έχουν ασκήσει μεγάλες πιέσεις στο πώς εκτελούνται δαπάνες βάσει του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση που θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο αργότερα φέτος, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς τη χρονική στιγμή. Μάλλον στο δεύτερο έμιση τη φετινής χρονιάς. Η αναθεώρηση αυτή θα εξετάσει τις προτεραιότητες, το που θα πρέπει να οδεύσει στο μέλλον ο ευρωπαϊκός προπολογισμός και επίσης θα υπάρξει συζήτηση για τα ζητήματα που τώρα μας απασχολούν στην πολιτική επικαιρότητα. Για να αναφέρω μεταξύ άλλων ως παραδείγματα την κρίση των προσφύγων και ούτω καθεξής. Το μήνυμα για την κοινή αγροτική πολιτική στο τρέχον πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αρκετά καθησυχαστικό, διότι τα χαρτοφυλάκια που έχουν ήδη προβλεφθεί για τα κράτη-μέλη δεν θα αγγιχθούν, δεν θα συζητηθούν. Και αυτό είναι συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το τρέχον πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε δεν θα υπάρξει αναδιανομή συγγνώμη, στον τίτλο 2 ε, για τα γεωργικά κονδύλια και δεν θα κατευθυνθούν προ άλλου άλλα κεφάλαια. Η σημασία του μηνύματος αυτού είναι ότι μπορούμε να, να ελπίζουμε σε κάποια σταθερότητα. Είμαστε σε φάση υλοποίηση των πολιτικών που έχουν αποφασιστεί, οπότε το μήνυμα που θα προκύψει από αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση είναι ένα μήνυμα καθησυχαστικό για το συγκεκριμένο τομέα. Επίσης θα κοιτάξουμε και κάποια ποιοτικά στοιχεία στις δαπάνες των τίτλο το ανέφεραν κάποιοι συναδελφοί σας, η κλιματική ευθυγράμμιση και η βιοπικιλότητα, η προστασία της είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20% του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού έχουν στοχευθεί και έχουν ε, εντοπιστεί για να επιδιωχθούν οι στόχοι αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Η πολιτική μας για το κλίμα είναι βεβαίως μέλος, μέρος όλου αυτού του 20% και θα είναι σημαντικό με την ανακοίνωση που θα προκύψει να σας δείξουμε ότι υπάρχει αποτελεσματική και σωστή χρήση των κομπηλίων της γεωργικής πολιτικής. Επίσης θα γίνει συζήτηση γενικότερη του προπολογισμού που θα επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, ιδίως όπως έχουν ε, υποχρεώσει εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και διαδικασίε απαλλαγή του κοινού προπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε ότι αποτελέσματα επιτυγχάνονται χάρη στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην ξεχνάμε ότι στη συζήτηση αυτή θα ενταχθεί και ε, το θεματολόγιο της απλούστευσης του Επιτρόπου Χόγκαν προκειμένου να αναζητήσουμε τρόπους να ξεφύγουμε από το μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος στην κοινή αγροτική πολιτική ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές μας αποφάσεις για το 2013 όπως είχαν τότε καθοριστεί οι μεταρρυθμίσεις. Θα υπάρξουν κάποιες κατεξουσοδότες και εφαρμοστικές πράξεις, γνωρίζετε τι θα ισχύσει εδώ, όμως επίσης αυτό είναι το σχέδιο της Επιτροπής. Θα δούμε τι προσπάθειες θα χρειαστούν στα πλαίσια της ενδιάμενης ε, αναθεώρησης, διότι θα εξεταστούν μελλοντικά όλες οι περιοχές δαπανών, όχι μόνο οι γεωργικές. Τέλος, έχει γίνει σαφές από τη συζήτηση σήμερα, αλλά το επισημάνω κι εγώ, η ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση σχετίζεται με μια πρόταση που στα τέλη του 17 θα πρέπει να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που μετά θα συζητηθεί στις αρχές του 2018. Θα τεθούν γενικότερα ερωτήματα για τις πολιτικές μας, όχι μόνο για την κοινή αγροτική πολιτική, για όλες τις πολιτικές που ενέχουν τα πάνες. Θα εντοπιστούν οι σχετικές και θα γίνουν οι σχετικές πολιτικές συζητήσεις και ένα νέο πλαίσιο θα αποφασιστεί για την περίοδο 2021-2028. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά ποιε είναι οι σχέσει, κύριε Διευθυντά, μεταξύ τη κοινή γεωρικής πολιτική και των εθνικών φακέρων, των εθνικών κονδυλίων γιατί μερικές φορές είναι μονόδρομος, μονοσήμαντη η κατέθεση. Πολύ σημαντικό το θέμα, κατάσταση στη Γεωργία και ξέρουμε ότι θα έχουμε μαζικές διαμαρτυρίες ε, γεωργών και το περιμένουμε αυτό. Γιατί συνεχώς μιλάμε για τις προκλήσεις και συμφωνώ με τον κύριο Γιάρο ότι θα πρέπει να επιλύσουμε και την τρέχουσα κατάσταση, την κρίση, να επιφέρουμε μια σταθεροποίηση τώρα και να μην περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί για το μέλλον εύκολο γίνεται συζητήσει. Το θέμα είναι πώ θα λύσουμε τα τωρινά προβλήματα. Τα τρέχοντα προβλήματα. Πρώτα να λύσουμε τα τρέχοντα προβλήματα και μετά να συζητήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι εμείς ε, Είμαστε πεπισμένοι για τη σημασία της γεωργίας, αλλά θα πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπους, τους υπουργούς, ε, τους συναδέλφους, τις πολιτικές ομάδες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρόσφερο κλίμα για τη γεωργία. Και επίσης να πούμε στους γεωργούς ότι δεν χρειάζεται να έρχονται σε εμά, γιατί είναι προφανές ότι εμείς ε, υποστηρίζουμε τα συμφέροντά τους. Θα πρέπει να κάνουν διαβήματα και προς ε, άλλους ευρωβουλευτές, σε άλλες επιτροπές. Επίσης δεν είναι μόνο θέμα κοινή γεωρική πολιτική, είναι το κλίμα, είναι η, η Δεν είναι μόνο η γεωργία αμυγός. Έχουμε και περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανάπτυξη και έχουμε και τους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν είναι αυτόνομη η γεωργία. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στις παγκόσμιες αγορές γιατί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία εξαρτάται και από την κατάσταση στην παγκόσμια γεωργία. Πρέπει να δούμε τι τάσεις υπάρχουν στην παραγωγή, πώς θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια. Και μεγάλες χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, πώς θα, θα δρομολογήσουν την παραγωγή τους. Και το θέμα είναι να αναπτυχθεί η γεωργία μας, όχι να, στην καταστρο... να οδηγηθεί στην καταστροφή. Γιατί έτσι θα χάσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο της γεωργίας. Ε, πρέπει να δείξουμε πυγμή λοιπόν κύριε Γιάρ κατά την πρόσπιση των θέσεων μας. Μέχρι τις 29 Απριλίου μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας αγαπητοί συνάδελφοι στις 12 το μεσημέρι. Δεν ξέρω κύριε Σιγητά, θα ξαναθέλατε το λόγο κύριε Γιάννα, αλλά σύντομα παρακαλώ. Σύντομα δύο παρατηρήσεις. Ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Η έκθεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, γι' αυτό περιμένω και την επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Θα δούμε εκεί πέρα τις τροπολογίες. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, η εξελίξη στην Ήπεθρο, το μποϊκοτάζ της ε, Ρωσίας, ε, μπορούμε όλα αυτά νομίζω να τα δούμε. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε στο θέμα μας. Κοιτάξτε, τα πρώτα πέντε σημεία ε, κάνουμε, στα πρώτα πέντε σημεία κάνουμε διαφήμιση της γεωργίας για να πείσουμε τους άλλους συναδέλφους μας εδώ μέσα. Να τους εξηγήσουμε ποια είναι η κοινή γεωργική πολιτική, να τους πούμε πως δεν είμαστε βαρέλοι χωρίς πάτο, είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και είναι νομίζω θετικό αυτό για τους συναδέλφους ε, στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού ακριβώς για να εξηγήσουν, ε, να εξηγήσουμε κι εμείς την πολιτική της Γεωργίας. Θυσίασα όπως σας είπα πέντε σημεία για αυτό το θέμα. Υπάρχουν όπως είπαμε και παράματα τα οποία δεν κοστίζουν, μείωση της γραφειοκρατίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και εκνευρίζει και τους γεωργούς και τους πάντες και τους επιβαρύνει. το άλλο που είπα χθε. συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Δηλαδή ποια θα είναι η μελλοντική γεωργική πολιτική. Ε, πολλοί συνάδελφοι έχουν πολλές ιδέες, αλλά δεν ήθελα τώρα να τα βάλω σε αυτή την έκθεση, γιατί δεν φτάνει και ο χρόνος και απευθύνω ξανά το ερώτημα προς τον Πρόεδρο τους ε, συντονιστέ. δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα μία συζήτηση. Ποια θα είναι η μελλοντική γεωργική πολιτική αλλά αυτό θα απαιτεί πολύ χρόνο. Δηλαδή, να ξεκινήσει τώρα, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, συναδέλφους να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε λίγο εδώ μέσα σε αυτή την έκθεση. Αλλιώς οι υπόλοιποι βουλευτές στο υπόλοιπο κοινοβούλιο θα μας διαλύσουν. Δεν ξέρω αν έχει και κάποια ιδέα ο πρόεδρο για το πώ θα γίνει αυτή η γενικότερη συζήτηση την οποία είπαμε. Γιατί νομίζω πρέπει να στείλουμε τώρα ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή Προπολογισμού ότι ξέρουμε τι θέμε και να είναι και ρεαλιστικό, έτσι. Γιατί εντάξει μπορούμε να λέμε ότι θέμε αυτά, να είμαστε χαρούμενοι μεταξύ μας, αλλά δεν θα, το, δεν μας τα δώσουν οι υπόλοιποι. Αυτά σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αστεριζόμαστε τις απόψεις σας, είμαστε στο πλευρό σας και έχουμε τη Δευτέρα στις 3 ε, ε, νέα συνεδρίαση με δημόσια κρόση. Παρακαλώ να είστε παρόντες. Αυτά με την δημόσια συνεδρίαση. Μία δίλεπτη τεχνική παύση, ένα σύντομο τεχνικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά επανερχόμαστε για τις συνεδρίες των συντονιστών και